Pan Przewodniczący! Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy, kolegów. E, Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλώς ήρθατε. Κυρίσω την έναρξη λοιπόν της ε, Συνόδου, πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, αφορά τη συζήτηση, την κοινή συζήτηση όσον αφορά τον προπολογισμό του 2012. Πρόκειται περί εκθέσεως της κυρίας Μπαλτζάνη και του κυρίου Φερνάντες η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 2012 ως τροποποιήθηκε το Συμβούλιο καθώς και έκθεση του κυρίου Μπέκερ για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Πηγαίνουμε λοιπόν στη συζήτηση. Η συνάδελφός μας, η Φραντσέσκα Μπαλτζάνη, θα ξεκινήσει τη συζήτηση. Είναι η συγγήτρια όσον αφορά αυτή την έκθεση. Κυρία Μπαλτζάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζούμε στιγμές κρίσης και αυτή η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι και κρίση εμπιστοσύνη. Κρίση εμπιστοσύνη που πλήττει όλου.